ο κύριος Μπρεζίνα. Είναι παρόν ο κύριος Μπρεζίνα. Eh, Καταψήφισα την έκθεση Μπέγκε για την eh, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι η προσέγγιση δεν είναι συστηματική ε, είναι άνευ το ποσό που δίνουμε κατά κεφαλή μετά από το αίτημα της Αυστρίας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν απολυθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις πραγματικές οικονομικές ανάγκες και το οικονομικό πλαίσιο. Αυτό όμως δεν γίνεται. Η προσέγγιση είναι εντελώς τυχαία και αυθαίρετη και επομένως πιστεύω ότι θα πρέπει να καθορίσουμε πολύ αυστηρά κριτήρια για την κινητοποίηση του Ταμείου. Γιατί τα κονδύλια τα οποία κινητοποιούνται έτσι δεν βοηθάνε. Θα είναι μόνο μια σπατάλη πόρων. Ευχαριστώ. Στο ψήφισμα για τις προοπτικές της αναπτυξιακής ατζέντα της Δόχα μετά την 7η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ, ο κύριος Καμάλ έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να εξηγήσω τη θέση μου σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ο λόγος για τον οποίο Πολλοί από εμά ενδιαφερόμαστε για τα θέματα του εμπορίου είναι για να βοηθήσουμε αυτού οι οποίοι βρίσκονται στι φτωχότερε χώρε του κόσμου για να μπορέσουν να εξέλθουν από την ένδια. Ένα από του καλύτερου τρόπου να το κάνουμε αυτό είναι να βοηθήσουμε του επιχειρηματίε στι μικρέ χώρε. Οι επιχειρηματίε <clears throat> είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν τη βοήθειά μα και είναι απαραίτητο να του υποστηρίξουμε. Θα πρέπει όμω να κοιτάξουμε και μέσα στα δικά μα σύνορα για να εξασφαλίσουμε ότι θα άρουμε του φραγμού για να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία σε εμπορικό επίπεδο με τι φτωχέ χώρε. Οι μικρέ χώρε στον κόσμο, οι φτωχέ χώρε θεωρούν ότι το εμπόριο είναι άνισο ει βάρο του. Εις βάρος βλέπουν τα διπλά στάνταρτ, τα φυτοϊγειονομικά, βλέπουν τις, ε, τους περιορισμούς που υπάρχουν, τις επιδοτήσεις για τις ε, αγροτικές εξαγωγές. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι με το εμπόριο εμείς βοηθούμε τις φτωχές χώρες να εξαλείψουν ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο. Ε? Κύριε Ντέβα, έχετε το λόγο, ναι. You have the floor, Mr. Deva. Come on. Μα έχετε το λόγο, κύριε Ντέβα, ορίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αν θέλουμε να ανακουφίσουμε την φτώχεια και την ανέχεια στον κόσμο πρέπει να αυξηθεί το παγκόσμιο εμπόριο. Αν όμω ακολουθήσουμε την οδό του προστατευτισμού, την κατοφερή οδό του προστατευτισμού, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να καθυστερήσουμε την καταπολέμηση της φτώχεια σε εκατομμύρια ανθρώπους που θα αποθάνουν. Και αν δεν αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή από τώρα και δεν προβλέψουμε το μέλλον μετά την κρίση τότε η κληρονομιά που θα αφήσουμε θα είναι τρομακτική. Δισεκατομμύρια άνθρωποι θα είναι, δεν θα είναι σε θέση να επιβιώσουν και οι εκκληματολογικές αλλαγές, η θέρμανση του πλανήτη και τέτοιου είδους καταστροφές θα χειροτερέψουν. Χρειάζονται τη βοήθειά μας και ο μόνος τρόπος να τους βοηθήσουμε είναι να αυξηθεί το παγκόσμιο εμπόριο και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο νέος υποψήφιος ε, Επίτροπος Εμπορίου με ακούει. Γράφεται ως επεξήγηση ψήφου προφανώς. Ο κύριος έχει το Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου αντίθετα από την άποψη του προηγουμένου ομιλητή είναι για μένα αντίθετη η άποψή μου. Δεν πιστεύω ότι το παγκόσμιο εμπόριο θα μπορέσει να βοηθήσει το ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων που ζουν σε γεωργία επιβίωσης να βγουν από την ένδια και την πείνα. Δεν είναι το παγκόσμιο εμπόριο. Η τροπολογία η οποία αναφέρεται στις δημόσιες υπηρεσίες και την ανάγκη οι να μπορέσουν να διατηρήσουν τον έλεγχο των δημοσίων ε, εταιριών, όπως είναι η υδροδότηση, η ενέργεια και όλα αυτά, που για μένα κεφαλαιώδης. Επειδή απερίφθη αυτή η τροπολογία, εγώ αναγκάστηκα να καταψηφίσω στο συνολικό ψήφισμα. Ευχαριστώ.